Ξεκινάμε με τον κύριο Άλιστερ. Μόνο μία επεξήγηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε τον λόγο για να εξηγήσετε το πώς ψηφίσατε στην εκθεσή Καζάκα. Ευχαριστώ. Κάθε μέρα όλο και περισσότεροι ψηφοφόροι μου δεν μπορούν πλέον να τα βγάλουν πέρα. Και μετά έχουμε μια τέτοια έκθεση εδώ πέρα και ανακαλύπτω πως 1,6 δις από τα χρήματα των Ευρωπαίων φορολογουμένων ξοδεύτηκαν σε αυτό το κτίριο. Και μετά ανακαλύπτω 9,3 εκατομμύρια δόθηκε στα πολιτικά κόμματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και μετά βλέπω πως επαναλαμβάνεται η δέσμευση για μείωση κατά 30% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2020, αλλά δεν γίνεται ούτε μία αναφορά στην πιο εξωφρενική εκπομπή όλων. Αυτή δηλαδή προκύπτει από την άχρηστη μετάβασή μας εδώ πέρα 12 φορές το έτος. Πρόκειται για μια έκθεση ανατριχιαστική σε σχέση με το όσα αποκαλύπτει για τη συμπεριφορά του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Άλιστερ. Κυρία Σίνοτ, για το ίδιο ζήτημα, έκθεση Καζάκα. Κύριε Σκόρμπετ, ναι. λοιπόν, ευχαριστώ Πρόεδρε. Να θέσω το σωστό πλαίσιο για τα σχόλια του κ. Άλιστερ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κοστίζει σε κάθε πολίτη 1,74 λίρες, λέω λίρες για τον κύριο Άλιστερ, το έτος. Εν συγκρίση, η Βουλή των Κοινοτήτων κοστίζει κάθε έναν Βρετανό πολίτη 5,75 λίρες ανά έτος. Η Βουλή των Λόρδων 1,77 ε, λίρα για κάθε πολίτη του Ηνωμένου Βασιλείου. Με άλλα λόγια, αυτό το κοινοβούλιο είναι πολύ φθηνότερο όσον αφορά τη λειτουργία του ανά πολίτη. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να επαναπαυθούμε στις δάφνες μας. Βεβαίως πρέπει να επαγρυπνούμε, πρέπει να περικόπτουμε τις δαπάνες. Και το επιχείρημα του κυρίου Άλιστερ περί των 12 ολομελιών το χρόνο που κοστίζουν τόσα χρήματα στο Στρασβούργο είναι βεβαίως μια σωστή παρατήρηση. Αλλά αυτή η απόφαση ε, δεν εναπόκειται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι απόφαση που αφορά τα κράτη-μέλη, που δυστυχώ στο Εδιμβούργο υπό την προεδρία του John Major κατέστησαν υποχρέωση για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, νομική υποχρέωση να ερχόμαστε εδώ 12 φορέ το χρόνο. Λοιπόν, καλό τα κράτη-μέλη να επανεξετάσουν αυτή την απόφαση. Ευχαριστώ. Κύριε Κόρμπετ, συνεχίστε με τι υπόλοιπε για Την έκθεση Σόντεργαρτ, για παράδειγμα. Okay. Εντάξει, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όχι, Αστρίτ, κάθισε κάτω. Κύριε Κόρμπετ, παρακαλώ. Λοιπόν, για την απαλλαγή του Συμβουλίου. Τι είστε πάλι σε αυτή η συμφωνία κυρίων που ήταν πριν από την άμεση εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ότι δηλαδή το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν την πλήρη ευθύνη ε, εσωτερικά για τον προπολογισμό τους, χωρίς ο ένας να μπαίνει στα χωράφια του άλλου. Ε, πρέπει να εξετάσουμε ξανά αυτή τη συμφωνία κυρίων, γιατί πλέον ο προπολογισμό του Συμβουλίου δεν αφορά μόνο την διοίκηση του συνομοθετικού αυτού οργάνου, αλλά και έναν προπολογισμό που θα αυξηθεί στο μέλλον για εκτελεστικές λειτουργίες στον τομέα της ΚΕΠΑ. Η συμφωνία αυτή κυρίων ποτέ δεν θα αφορούσε εκτελεστικές λειτουργίες, ποτέ δεν θα εξαιρούνταν αυτές από την κοινοβουλευτική εξέταση και πρέπει λοιπόν να ξεκινήσουν συζητήσεις για αυτή τη συμφωνία κυρίων. Έχει τον λόγο για την έκθεση Καζάκα. Euh, Κύριε Πρόεδρε, έχω απόσχει από την ψηφορία την απαλλαγή 2007 για το προϋπολογισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω κάποιων παραγράφων της εκθέσεως αυτής που εμπνέονται από παραπληροφόρηση και από αναλήθειες που διαδίδονται μέσω των μέσων ενημέρωσης και εδώ όσον αφορά το επικουρικό συνταξιωτικό ταμείο των μέλων και ο Σκονμπέντιτ μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος 40 χρόνια εισφορών δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί για να ταξιδοτηθούν οι, τα πρώην μέλη και οι χείρε του κλπ. Λοιπόν, αν θεωρεί ότι οι βουλευτέ, τα μέλη του Συνταξιωτικού τομείου, του Επικουρικού Συνταξιωτικού τομείου δεν πρέπει να συμμετέχουν στην ψηφοφορία για την απαλλαγή, καλά θα έκανε ε, να καθαρίσει τα του οίκου του πρώτα. Εξάλλου, συμμετέχει στι ε, ψηφοφορίε τη πτώση του προπολογισμού μα που χρηματοδοτούν τι αποζημιώσει του και τι αμοιβέ του. Ε, λόγω διαφανείας ε, επί πέντε χρόνια μία φορά πάτησε σε μία συνεδρίαση μιας ε, επιτροπής της οποίας είναι μέλος. Λοιπόν, εδώ στο νομοθετικό μας έργο δεν αξίζει εδώ να κάνουμε συνεντεύξεις τύπου και να φωνασκούμε. Χρειάζεται περισσότερη διακριτικότητα. Αλλά σαν πρώην ε, φοιτητής του 68 δεν μπορούσε να περιμένει κανείς τίποτα παραπάνω από αυτόν. Και οι δηλώσεις εδώ ακόμα και αν προέρχονται από τους προέδρους των ομάδων δεν θα αλλάσουν ε, επουδενή τις νομικές ευθύνες αυτού του κοινοβουλίου που είναι γραμμένες ε, στο μοσαϊκό νόμο αν θέλετε. Ε, Τώρα, για την έκθεση Φιέλνερ, ο κ. Κάλαχαν, που επίσης έχει ζητήσει να δώσει μια διευκρίνηση για την έκθεση Τικάου και άλλη μια επεξήγηση για την έκθεση Α, δεν είναι εδώ. Mm. Οκ. Ωραία. Το κλείσαμε αυτό. Έκθεση Φιέλνερ. Κύριος Χάναν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μόλις υπερψηφίσαμε τη χρηματοδότηση για πάρα πολλές αποκεντρωμένες υπηρεσίε φαρμάκων, εξωτερικών συνόρων, ε, ποια είναι τα άλλα εκεί, ασφάλεια της αεροπορίας κτλ. Έχω αντίρρηση για τρει λόγου. Υπάρχει το ευρωσκεπτιστικό επιχείρημα, το δημοκρατικό και το νομικό. Το ευρωσκεπτιστικό τώρα δεν. βεβαίω βεβαίως αναμένω να τύχει στήριξη. Δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα να γίνονται σε επίπεδο των Βρυξελών. Νομικό επιχείρημα. Α, όλες αυτές οι υπηρεσίες θα είχαν νομική ισχύ αν είχε περάσει η συνθήκη της Λισαβόνας. Αυτή τη στιγμή δεν έχουν. Το δημοκρατικό επιχείρημα όμως νομίζω ίσως να σταθεί ακόμα και με τους φεντεραλιστές συναδέλφους. Όταν ένα κοινοβούλιο τέτοιο, όπως το δικό μας, δίνει υπεργολαβία εργασίες ε, σε αυτούς τους οργανισμούς και δεν τους βλέπουμε μετά ποτέ και μετά να μένουμε να ασκήσουν αυτή την πολιτική και εμείς απλά να υπογράφουμε τις επιταγές, έχουμε μειώσει την δημοκρατία μας. Ο Χάγεκ είπε πως η παραχώρηση εξουσίας είναι το πρώτο βήμα με το οποίο μια δημοκρατία παραδίδει τις εξουσίες της. Οι συνάδελφοι λοιπόν είτε είναι υπέρ είτε κατά της ομοσπονδιακής Ευρώπης να το ξέρουν. Τι είναι παιδίδας? Κυρία Σύρη, ε, έχει ζητήσει να κάνει πολλές επεξηγήσεις ψήφου. Παρακαλώ κάντε τη, στιγμή μετά την άλλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σύρι το μικρό μου όνομα. Μοβίρ λέγομαι στο επώνυμο. Ευχαριστώ πολύ. Έχω πράγματι αρκετέ εξηγήσει ψήφου, δεν το έχω κάνει αυτό στο παρελθόν, αλλά θεωρώ σημαντικό να το κάνω σήμερα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να αναφερθώ στην έκθεση Γκροστέτ, την οποία ψήφισα και υποστήριξα και τις προτάσεις της Επιτροπής Μεταφορών, γιατί θεωρώ πως ε, δύο κανονισμοί που ασχολούνται με αυτό το θέμα πρέπει να γίνουν ένας ε, κανονισμός και είναι αυτό ένα βήμα δικαιολογημένο, ένα βήμα προς την δημοκρατία και μείωση του διοικητικού άχθους. Μετά αφαιρθώ στην εκθεσικός και αυτή την υποστήριξα γιατί και αυτή μας βοηθάει να γίνει πιο συνεπής αυτός ο κανονισμός, ιδιαίτερα δεδομένη της διεθνούς φύσης ε, του αντικειμένου. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε την δυνατότητα να έχουμε πανευρωπαϊκές έρευνες στα αρχεία για να προστατευτούν με αυτόν τον τρόπο οι πελάτες μας έναντι αθέμη του ανταγωνισμού. Κατόπιν έκθεση Γκρόσερ. Και αυτή την υποστήριξα γιατί και αυτή είναι αφιερωμένη σε ζητήματα μεταφορών και θα βελτιωθεί έτσι η επιτελεσματικότητα της εσωτερικής αγοράς, θα μειωθεί το διοικητικό κόστος και θα επιτρέψει δικαιότερο ανταγωνισμό. Κατά την άποψή μου για να ολοκληρωθεί η ε, κοινή αγορά στην Ευρώπη πρέπει να έρθουν και οι περιορισμοί στις εσωτερικές αγορές των κρατών μελών στο προσχέσμελο. Η άλλη έκθεση για την ενεργειακή αποτελεσματικότητα των κτηρίων και αυτή την υποστήριξα γιατί υπάρχουν πραγματικά προκλήσεις σε αυτόν τον τομέα. Μπορούμε να εξοικονομήσουμε 20% της κατανάλωσης ενέργειας από την αποτελεσματική χρήση της. Όσον αφορά δε τις επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, αυτές βοηθούν και στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας, γιατί έτσι θα δημιουργήσουμε όσο δουλειέ δημιουργούμε και με τις παραδοσιακές επενδύσεις και ίσως και περισσότερες και έτσι θα επιτύχουμε τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα έτσι θα βγούμε και από την κρίση θα δημιουργήσουν περισσότερες θέσεις εργασίας και θα μειωθεί η εξάρτησή μας από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Τώρα, η έκθεση κορός που αφορά τους οργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας και αυτήν την υποστήριξα γιατί τα προβλήματα σε αυτόν τον τομέα ειδικά όσον αφορά την επίβλεψη ε, συνεισέφεραν και αυτά στην παγκοσμία οικονομική κρίση. Ε, τομέας ε, δραστηριοποίησης αυτών των υπηρεσιών είναι μεν παγκοσμίω, αλλά βρίσκονται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε δεν ξέρω αν είναι αποτελεσματική εδώ η ευρωπαϊκή νομοθεσία για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους. Για να το ξεπεράσουμε αυτό λοιπόν πρέπει να συνεργαστούμε με τρίτες χώρες. Τώρα η έκθεση αφορούσε τα δικαιώματα των επιβατών σαλάσιες ε, ε, και γενικά στις πλωτές μεταφορές. Είναι ένα πολύ καλό βήμα, αυξάνονται τα δικαιώματα των επιβατών και αυξάνονται τα ίσα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες για τους ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτά τα μέσα μεταφοράς. Η έκθεση Αλμπερτίνη που αφορά τα δικαιώματα επιβατών σε λεωφορεία και πούλμαν. Και αυτή την υποστήριξα. Γιατί τα μέτρα αυτά τελικά θα βοηθήσουν στην εξάλληψη της αδικίας, της ανισότητας στην Ευρώπη που ίσχυε μέχρι στιγμής ε, κάτι το οποίο συμβαίνει ήδη σε αεροπορικές μεταφορές και στις σιδηροδρομικές μεταφορές και τα δικαιώματα των επιβατών. Επειδή δε αυτό σχετίζεται και με εταιρείε ε, με νέες εταιρείε οι οποίες αντιμετωπίζουν και νέες ε, ε, υποχρεώσεις πρέπει να τους δοθεί μια μεταβατική περίοδος. Τώρα η επόμενη έκθεση για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών. Τα συστήματα αυτά έχουν αποδείξει την αποτελεσματικότητά τους, έχουν κάνει τις μεταφορές πιο ασφαλείς, έχουν επίσης συνεισφέρει στο να επιτύχουμε έναν πολιτικό στόχο, δηλαδή να γίνουν οι μεταφορές πιο καθαρές. Γι' αυτό υπερψήφισα και αυτή την έκθεση. Η έκθεση Στόκμαν, το δεύτερο πρόγραμμα Μάρκο Πόλο δηλαδή, πρέπει πράγματι να υποστηριχθεί γιατί στο πλαίσιο αυτό θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα μποτιλιαρίσματα, να βελτιώσουμε τα περιβαλλοντικά μέτρα και την χρήση συνδυασμένων μεταφορών. Ανησυχώ όμως για το ότι κάθε χρόνο οι αιτήσει για οικονομική ενίσχυση και ο αριθμός των έργων που χρηματοδοτούνται με αυτά τα κονδυλία μειώνεται χρόνο με το χρόνο. Τώρα, για την έκθεση της ΣΑΜ, την οποία υποστήριξα, ε, την υποστήριξα γιατί οι σιδηροδρομικές μεταφορές είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο μεταφορών ακόμα και σήμερα παρά την μείωση των εμπορευματικών μεταφορών ε, μέσω σιδηροδρόμου. Συμφωνώ με τον εισηγητή δε πως αυτό το νομοθέτημα πρέπει να προετοιμαστεί κατά τρόπον ώστε η σιδηρόδρομη θα είναι αποτελεσματική για όλους τους χρήστες στο μέλλον. Σήμερα το πρωί συζητήσαμε τις εκθέσεις που ήταν μέρος του πακέτου υγείας και ψηφίσαμε και την έκθεση για τα δικαιώματα των ασθενών έκθεση στην διασυνοριακή παροχή υγείας έκθεση την οποία επίσης υποστήριξε γιατί θεωρώ πως εδώ και πάρα πολύ καιρό οι βουλευτές ήταν ικανοποιημένοι με το να νομοθετούν εδώ οι νομικοί. Εγώ νομίζω πως πρέπει να νομοθετούν οι πολιτικοί, οι αιρετοί εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών. Έχει φτάσει η ώρα να ε, υιοθετήσουμε πια αυτή την οδηγία. Τώρα, η έκθεση Τρακατέλη για τις σπάνιες ασθένειες είναι συνέχεια του θέματος των δικαιωμάτων των ασθενών και αυτή την υποστήριξα, αλλά δεν υποστήριξα την τροπολογία υπαριθμών 15. Αυτό είναι θέμα του προηγούμενου αιώνα. Η πολιτική δεν πρέπει να μπαίνει στα πόδια της γενετικής έρευνας. Τώρα η έκθεση για την ε, κινητικότητα στις πόλεις ε, την υπερψήφισα γιατί παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μεταφορά επιφατών και αγαθών οπότε έχει φτάσει η ώρα να γίνει μια ξεχωριστή στρατηγική και για αυτό το θέμα. Και τέλος θα ήθελα να αναφέρω την έκθεση της κυρίας Γένσεν για τα έξυπνα συστήματα μεταφορών και το σχέδιο δράσης επειδή ε, έχει στο κέντρο την συνεργασία, την τυποποίηση, θεωρώ πως και αυτή η έκθεση ήταν αναγκαία και πρέπει να την υπερψήσω. Ευχαριστώ. Κύριε Χάνεν, ε, ε, έχετε και μια δεύτερη επεξήγηση. Να σας ακούσουμε για, τις, για την εκτίμηση επιστολικής ικανότητας. Σήμερα γιορτάζουμε την, τη γέννηση του εθνικού μας ποιητή. Είναι επέτειος των του μεγαλύτερου Άγγλου και δραματουργού που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότης. Είναι χαρακτηριστικό το έργο του Σέξπιρ ότι οποιαδήποτε εμπειρία α, απεικονίζουμε εκεί, α, φωτίζονται πιο πολλοί εμπειρίες εκεί στα έργα του από ό,τι στη ζωή μας. Ο, κύριος Τζον Κωστά είναι από το Ριχάρτο δεύτερο αναφέρονται τα προβλήματα τα δημοσιονομικά της Βρετανίας και της καταστάσεως στην ε, Ευρώπη. Αυτή η γη τόσων αγαπητών ψυχών, αυτή η αγαπητή γη έχει νοικιαστεί σαν να είναι ένα κτίριο. Ακούστε την περιγραφή τόσον αφορά τη συνθήκη της Λισαβόνα ή το Ευρωπαϊκό Σύνταγμα. Η Αγγλία που δεσμεύεται από τη θάλασσα σκάνε τα κύματα στην παραλία. Η Αγγλία τώρα έχει δεσμευτεί και τη χτυπάνε, τα χρέη και η γραφειοκρατία. Αυτή η Αγγλία που ήθελε να κατακτήσει άλλους τελικά αυτοκατακτήθηκε με ντροπή. Λοιπόν, να υπάρχει καλύτερη ερμηνεία από αυτή, περιμένω να την ακούσω. ¿eh? Δεν ήξερα ότι ήσασταν ραψοδός. Ο κύριος Καμάλ για την έκθεση Τικάου, για τα κτίρια. Uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα να μιλήσω. Όταν ψηφίζουμε θέματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι όταν ψηφίζουμε ένα θέμα θα πρέπει να ηγούμεθα ηθικώς. Είναι σωστό εμείς να μιλάμε για ενεργειακή αποδοτικότητα. Εγώ ειλικρινά δεν έχω κανένα πρόβλημα να γίνει κάτι σε ευρωπαϊκό, εθνικό ή τοπικό επίπεδο αλλά νομίζω ότι μπορούν να γίνουν περισσότερα σε τοπικό επίπεδο, αλλά είναι καλό να μοιραζόμαστε τι βέλτιστε πρακτικέ και ιδέε σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Όμω, ηγούμενοι θα πρέπει να ηγούμεθα και ηθικώ. Πώ μπορούμε να μιλάμε για ενεργειακή αποδοτικότητα των κτηρίων, όταν εμεί συνεχίζουμε να έχουμε δύο αίθουσε για το Κοινοβούλιο, μία στο Στρασβούργο και μία στι Βρυξέλλε. Και τι γίνεται αν σε εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο του Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο όταν μιλάμε για δεκάδε. χιλιάδε τόνου εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακο κάθε χρόνο. Ήρθε η ώρα να σταματήσουμε την υποκρισία, να ηγηθούμε και να κλείσουμε το Κοινοβούλιο του Στρασβούργου. Κύριε Καμάλ, ε, θέλετε να εξηγήσετε την ψήφο σα και για την έκθεση Μπόη, έτσι δεν είναι. Θα ήθελα να ξεκινήσω και εγώ δίνοντα χαρακτηρία στον Τζον Μπόβις και του ευχόμαστε όλοι καλή ανάρρωση και ευτυχώ εκείνο μπόρεσε να εκμεταλλευτεί το σύστημα υγεία μια άλλη χώρα. Βρετανό ον εκμεταλλεύτηκε τις υπηρεσίες υγείας του Βελγίου. Και βεβαίως αυτό αποτελεί ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Δηλαδή όλοι οι πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση θα μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις για το πού θα ε, πάνε για τις υπηρεσίες ε, υγείας. Εάν δείτε τους ε, ρυθμούς ανάρρωσης ανάλογα με τις διάφορες ασθένειες διάφορες χώρες, είναι ένα στοιχείο το οποίο θα επιτρέψει στους ε, ασθενείς να επιλέξουν πού θα αναρρώσουν καλύτερα και να εκμεταλλευτούν εκεί αυτές τις υπηρεσίες υγείας. Είναι ένα θετικό βήμα. Βεβαίω συχνά εγώ ασκώ κριτική στις μας εδώ πέρα, αλλά νομίζω εδώ πως έχουμε ένα θετικό βήμα. Να προσφέρουμε δηλαδή μεγαλύτερη ποικιλία και επιλογή στους πολίτες της Ένωσης. Σας ευχαριστώ. Ωραία, κυρία Ρόιτοβα, έχει μία επεξήγηση για την έκθεση Καζάκα και άλλη μία για την έκθεση Κρόλη. Λόγω στην κυρία Ρόιτοβα. Κύριε Πρόεδρε, δεν υπερψήφισα την έκθεση Καζάκα η έκθεση αφορά το επικουρικό συνταξιδοτικό ταμείο των ε, βουλευτών και εγώ συνεισφέρω σε αυτό το ταμείο. Δεν θέλω να υπάρχει σύγκρουση ε, συμφερόντων και γι' αυτό έχω απόσχει από αυτή την ψηφοφορία. Και γι' αυτό στα πρακτικά της ε, Συνόδου παρακαλώ να σημειώσω ότι δεν υπερψήφισα την έκθεση Τρακατέλη για λόγους βιοηθικούς. Και μετά, Πρόεδρε, με ακούτε, ακούτε, να συνεχίσω. Η έκθεση Τρακατέλη. Μπορείτε να γράψετε στα πρακτικά ότι δεν το υπερψήφισα, δεν υπερψήφισα την έκθεση αυτή. Και τώρα επεξήγηση για την έκθεση Κράουλη. Καταψήφισα την έκθεση αυτή διότι δεν είναι ε, συνεπής, αλλά σε 40-50 χρόνια θα πρέπει να καλύπτονται τελικά τα πνευματικά δικαιώματα των ε, καλλιτεχνών. Χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία, χρειάζεται καλύτερη οργάνωση των ενώσεων των καλλιτεχνών που συλλέγουν τα δικαιώματα των καλλιτεχνών. Μελέτες συνεπιών δείχνουν ότι μόλις το 2% των εσόδων μοιράζεται στους καλλιτέχνες, τα υπόλοιπα χρήματα τα εισπράττουν οι δισκογραφικές εταιρείες και οι πιο δημοφιλείς καλλιτέχνες για τους νέους καλλιτέχνες πρέπει να κάνουμε κάτι και θα πρέπει να δούμε και τι γίνεται με τις δισκοθήκες, τις μεγάλες, τις βιβλιοθήκες, τις δανειστικές κλπ. Ε, δεν ήταν σωστά τα μέτρα από την Όταν γι' αυτό κατευθύνει την έκθεση. Η κυρία Φουρέ έχει επεξηγήσει ψήφου για την έκθεση Γέντσεν και για την έκθεση του Κυρία Φουρέ, έχετε το λόγο. Oui. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όσον αφορά την έκθεση Γιάνσεν, υπερψήφισα την έκθεση για την πρόταση οδηγίας όσον αφορά την ε, χρήση των ευφυών συστημάτων στις μεταφορές. Θέλουμε υπάρχει αντιδικότητα όσον αφορά τις επικοινωνίες και τεχνολογία της πληροφορικής στις μεταφορές. Η καινοτομία στον τομέα των μεταφορών θα πρέπει να ενθαρρυνθεί κυρίω όσον μπορεί να βελτιώσει, βελτιώσει την ασφάλεια των οχημάτων. Όμω η καινοτοπία χάνει τη χρησιμότητά τη αν δεν εγγυόμεθα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο. Αυτή η οδηγία θα πρέπει να επιτρέπει να συμβάλλουμε στη μείωση του αριθμού των θανάτων στου ευρωπαϊκού δρόμου, μειώνοντα ταυτόχρονα και τον κίνδυνο των συγκρούσεων και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων. Υπενθυμίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καθόρισε σαν στόχο να διαιρέσει στο ίμιση αριθμό των νεκρών στου δρόμου μέχρι το 2010, αν συγκρίσει με το επίπεδο του 2000. Όσον αφορά αυτό, λυπούμε διότι η οδηγία τη συνοριακή συνεργασία για την οδική ασφάλεια που ψηφίσαμε εδώ και αρκετού μήνε δεν έχει οθετηθεί πάντα από την Υπουργεία Μεταφορών τη Ευρωπαϊκή Ενώση, ότι θα επέτρεπε και εκεί να σωθούν ζωέ, διευκολύνοντα την επιβολή κυρώσεων κατά των οδηγών που κάνουν παραβάσεις άλλο κάτω μέλο από εκείνο στο οποίο είναι καταχωρημένο το όχημά του. Όσον αφορά τώρα την έκθεση του κύριου Τισάν, όσον αφορά το διάδρομο σιδηροδρομικών εμπορευματικών μεταφορών, θα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέτει σε αυτή την έκθεση όσον αφορά τα ευρωπαϊκά σιδηροδρομικά δίκτυα για ανταγωνιστικό εμπόριο, μεταφορά εμπορίου. Η περισσότερη την έκθεση επέτρεπε να βελτιωθεί ο, το μεταφορά εμπορευμάτων μέσω των σιδηροδρόμων. Μια ευρωπαϊκή δράση σε αυτό το τομέα είναι κάτι απαραίτητο. Η παρούσα λειτουργία τη μεταφορά εμπορευμάτων σιδηροδρόμου δεν είναι ικανοποιητική. Ε, πολύ λίγα εχέγγυα υπάρχουν όσον αφορά την αξιοπιστία των ωραρίων για τι επιχειρήσει εκείνε που θα χρησιμοποιήσουν του σιδηροδρόμου για να μεταφέρουν τα εμπορεύματά του. Λοιπόν, θα πρέπει τη μεταφορά εμπορευμάτων με του σιδηρόδρομο να τον κάνουμε πιο εικιστική για τι εταιρείε και θα πρέπει τελικά περισσότερα εμπορεύματα να πηγαίνουν μέσω στο δρόμο από ότι το δρόμο θα μειώσουμε εκπομπέ ε, διοξιδίου του άνθρακο και θα μειωθούν και συμφορεί στου δρόμου. Ελπίζω οι Υπουργοί Μεταφορών των κρατών μελών να ακολουθήσουν τον δρόμο που άνοιξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προ ένα ευρωπαϊκό σιδηροδρομικό δίκτυο το οποίο θα είναι πιο αποδοτικό. Και τώρα δίνω το λόγο όσον αφορά την έκθεση Τρακατέλη στον κύριο Πόσελτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ καταψήφισα την έκθεση Τρακατέλη λόγω της σκανδαλώδους τροπολογίας 15 που εξισώνει και μπερδεύει την ε, θεραπεία ασθενών με την ε, δολοφονία γέννητων ανθρώπων. Πλέον μιλάμε για ριζική αμφισβήτηση του δικαιώματος στην ζωή και δεν έχει δικαίωμα στη ζωή ένα αγέννητο παιδί μόνο και μόνο γιατί είναι άρρωστο. Πρόκειται περί δολοφονίας. Γι' αυτό είναι απαράδεκτη και η έκθεση Τρακατέλη και η τροπολογία αυτή είναι σκάνδαλο που επιβαρύνει το κοινοβούλιο μας, το οποίο πάντα είχε μεγάλες κατακτήσεις στο θέμα της βιοειθικής και την προστασία του εισαγέννητης ζωής. Ευχαριστούμε κύριε Πόσελτ για την έκθεση ΟΝΤΗ για τις εκτελεστικές υπηρεσίες. Κυρία Γκρέσλε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην ψηφοφορία για την απαλλαγή, για πρώτη φορά όσο καιρό είμαι βουλευτής, καταψήφισα την απαλλαγή της Κομισιόν. Και θέλω να εξηγήσω γιατί. Πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο η Κομισιόν ε, χειρίστηκε την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. Έχουμε πάρα πολλά προβλήματα, πολύ μεγάλη διαφθορά, πολλά ευρωπαϊκά χρήματα έχουν εξαφανιστεί. το 2008 μόλις ξεκίνησε να παγώνει τα κονδύλια η Κομισιόν, το 2007 χάσα πάρα πολλά λεφτά και δεν υπάρχουν συστήματα ελέγχου ή υπήρχαν συστήματα ελέγχου τα οποία λειτουργούσαν τελείως ατελώς στην Ρουμανία έχουμε πολύ μεγάλο ε, ποσοστό διαφθοράς ε, και δεν λειτουργεί σωστά η δικαιοσύνη. Θέλω λοιπόν να στείλω ένα μήνυμα και να πω και στην Κομισιόν πως στο μέλλον πρέπει να χειριστεί διαφορετικά τις διευρύνσεις και θα έπρεπε να παρακολουθεί τα πράγματα για να έχουμε καλύτερες επιτυχίες στο μέλλον. Εγώ θέλω να βοηθήσουμε την ε, Κομισιόν και να υπάρχουν συστήματα οικονομικού ελέγχου που θα είναι άξια του ονόματός τους. Διαφορετικά θα έχουμε ένα πρόβλημα διαρκές για ολόκληρη την Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Διακόπτουμε μέχρι τις 3.